άρθρο 30 παράγραφος 5 για τον σχηματισμό των ηλεκτρικών ομάδων έχουν δοθεί στον πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πω πως οι ε, γνωστοποιήσεις της εκλογής των μελών προβλέπονται στο άρθρο 183 θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Επίσης, τα μέλη τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την εκλογή τους θα πρέπει να δηλώσουν υπευθύνες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 πως ε, πριν καταλάβουν την ε, θέση τους σύμφωνα με το άρθρο 7 του ε, κανονισμού για την διεξαγωγή άμεσων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δηλώσουν πως δεν ασκούν καμία δραστηριότητα η οποία είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του Ευρωβουλευτή. Ε, όταν κάποιος κάνει αυτή τη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, μπορεί να καταλάβει την θέση του και να συμμετέχει με όλα τα δικαιώματα μέχρι να εξεταστεί αυτή η εντολή ή μέχρι κάποιος να προβάλλει κάποια αντίρρηση. Οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταθέσει αυτή τη δήλωση περί ασυμβίβαστου να το κάνουν άμεσα. Σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού μας, θα πρέπει να προχωρήσουμε